Πριν ε, ψηφίσουμε, να κάνω μια ανακοίνωση. Να σας πω ότι βάσει προηγούμενης απόφασης η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για το σχέδιο της διαδικασίας για το πρόσθετο πρωτόκολλο για τις εμπορικές ε, ε, διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ θα παραμείνει, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Επειδή 9 και 10 Ιουνίου είναι ε, προθεσμία για το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 11 Ιουνίου, 6 ε, το απόγευμα, στη δική μου ε, γνωμοδότηση. 11 Ιουνίου, 6 το απόγευμα. Πέρα των ανακοινώσεων λοιπόν, να περάσουμε στις ε, ψηφοφορίες για το σχέδιο ψηφίσματος, το οποίο κατέθεσε ο Μάριο Νταβίδ και ο κύριος Λάγκε για τις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύο τμήματα. Δεν είναι η συμφωνία αυτή καθεαυτή, ούτε ο κανονισμός. Είναι πρόταση ψηφίσματος, την οποία κατέθεσαν από κοινού οι εισηγητές ε, της ε, συνεδρικής διαδικτασίας και του κανονισμού για το θέμα αυτό. 83 τοπολογίες κατατέθησαν σε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε που ενοχλώ, έχω ξεχάσει την κάρτα μου όμως. Μπορώ να ψηφίζω δια ανατάσεως χειρός. Yeah, προσοχή παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα πολύ καλά την ανακοίνωσή σα για τη συμφωνία ΑΚΑ. Ε, είχα την εντύπωση ότι στην ε, συνεδρία των συντονιστών σήμερα το πρωί συζητήσαμε και ότι η άποψη όλων ήταν να προχωρήσουμε προς μια προφορική ερώτηση στην Ολομέλεια και να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε τα νομικά θέματα που συνδέονται με αυτή τη συμφωνία. Αυτή ήταν η συμφωνία των συντονιστών. Και εδώ εσείς μας λέτε για τροπολογίες και για ψηφοφορία. Τα έχω χάσει. Είτε έκανα λάθος, είτε... Αλλά βλέποντας και τον Ντανιέλ και άλλους, ε, άλλου είδους συμφωνία νομίζω είχαμε κάνει το πρωί. Όχι. Εγώ έθεξα αυτό το ερώτημα. Αλλά δεν με υποστήριξε κανείς. Και έτσι δεν υπήρξε αλλαγή. ο, χωρίς μικρόφωνο. Πέρα από το ECR υπήρξε σαφής υποστήριξη όλων των ομάδων να ακολουθήσουμε την σύσταση της γραμματείας. Τότε εγώ έκανα λάθος, λέει ο Πρόεδρος. And, uh, Όντως, όλοι οι υπόλοιποι συντονιστές ε, είχατε συμφωνήσει. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν. Λάθος δικό μου. Άρα πρέπει να αναβληθεί η προθεσμία. Στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών θα καταλήξουμε σε μια νέα προθεσμία. Ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Να ελέγξουμε καταρχάς, να δούμε αν έχουμε σωστό αριθμό εκπροσώπων από κάθε πολιτική ομάδα. Άρχεται η ψηφοφορία. Please, all, all, all of you should... Πιέστε ένα από τα δύο κουμπιά, όποιο θέλετε. Ε, Plus e Okay, it's okay. Including the vote. Εντάξει λοιπόν, συμπεριλαμβάνουμε και την ψήφα του συναδέλφου που δεν έχει την κάρτα του. Τροπολογία 31 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται να κάνουμε μια επαλήθευση. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 32. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 και πάλι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές να κάνουμε μια επαλήθευση γιατί δεν είμαι βέβαιος. Τρίτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη πληροφορία. Εγκρίνεται. 36. Κατά τμήματα και πάλι. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Συγγνώμη πίπτη. 38. Υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37. Ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 40 και 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 43 και 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40, θέλετε παλήθευση γιατί την 45, είστε βεβαίως. Όχι. 46, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 50. Κατά τμήματα. Τρία μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. Δεν είδα τι ψήφισε το Ελφ Ωραία. Επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. 50, δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is... Πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεν μέτρησα το έλκη γιατί δεν είδα τις ψήφους. Τρίτο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 56, απορρίπτεται, συγγνώμη, ο κύριος Σόλτ. Απορρίφθηκε με την τροπολογία, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι στην παράγραφο 10 λέει ότι, λέγεται ότι κανείς από τους πολίτες δεν έχει ενημερωθεί. Στην προηγούμενη εβδομάδα το συζητήσαμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια και υπήρχε κάτι το οποίο αφορούσε τα συνδικάτα. Ακόμα και αν έχουμε λοιπόν το θέμα αυτό, έχουμε τη συνεχή διαδικασία και χάνονται τα συνδικάτα και ήθελα να το θίξω το γεγονός αυτό. Αιτιολογήσατε λοιπόν την ε, τροπολογία σας. Η 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 και 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο κύριος Νταβίτ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους Ναι, προφορική τροπολογία θέλω να κάνω. Στην πρώτη τελευταία παράγραφο ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει αμέσως να συνδράμει την Κολομβία και το Περού. Μήπως θα έπρεπε να λέμε ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι διατεθειμένοι να συνδράμει, γιατί τι θα γίνει αν δεν του ζητήσει κανείς τη συνδρομή τους. Νομίζω ότι είναι πιο λογικό. Είναι προφορική τροπολογία, όχι είναι η συμβαστική τροπολογία του 14, στην παράγραφο 14. Δεν είχα την ευκαιρία να το θέσω, συμφωνείτε. Το να λέμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε, εφόσον μας ζητηθεί. για τη συμβιβαστική τροπολογία. Ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι έτοιμη να συνδράμει τη Κολομβία και το Περού. Υπάρχει κάποια έσταση για την προφορική τροπολογία, επομένω δεν έχουμε. Η συμβιβαστική τροπολογία 4 ως έχει υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 62 καταπίπτει, 64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 να ελέγξουμε το 7ο τμήμα. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για το 7ο τμήμα. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 65. Καταπίπτει. Περνάμε στην 68. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 κατά τμήματα το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τρίτο τμήμα υπέρ Επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Στο δεύτερο τμήμα λοιπόν έρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είδα τι ψήφισε το ΕΛΚ. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές να κάνουμε μια παλήθευση. 73 έρχεται η ψηφοφορία. 73. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 74. Καταπίπτει. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. το 76. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 και 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 και 80 όχι μόνο την 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, η 6 συγγνώμη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 και 8. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 10. Κατά τμήματα. Όχι, συγγνώμη, προφορική τροπολογία. Από τον Μπέρντ Λάγκε στην τροπολογία 10 Απλώ αντί για good να λέμε κούντ. Υπάρχει κάποια ένσταση. Όχι, ωραία. Να ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. απόχέ Απορρίπτεται. Επαλήθευση για την τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. And vote Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι 14 και 15 τώρα, που είναι ταυτόσιμες, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτονται. 16 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση για την 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Είμαστε στην 21, έτσι, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ. Και 28 μαζί. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 και με προφορική τροπολογία. Το έχετε στους φακέλους το κείμενο του Μπεντ Λάγκε. Υπάρχει κάποια ένσταση για την προφορική τροπολογία. Όχι, ωραία να ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση. Για την τροπολογία 30 με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. πέραση ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. εγκρίθηκε 20 ψήφοι υπέρ, του 21 υπέρ, 4 κατά, 3 αποχές, συγχαρητήρια στους δύο συνεισηγητές.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 δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το σφυρί μου, αλλά παρακαλώ. Okay. Item 14. Σημείο 14. Προσφόρηση Ευρωπαϊκή Ένωση στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος. Πρόκειται για ένα από τους πολλούς οργανισμούς ε, δασικών αγαθών, στους οποίους δεν έχει προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κυρία Μουσκαρδίνη είναι η εισηγήτρια που δεν βρίσκεται εδώ και θα αντικαταστήσει ο κύριος Κάσπαρη. Συντονιστές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ντάνιελ, έχει το λόγο για να μας κάνει την παρουσίαση του θέματος και να αρχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η συνάδελφος Μοσκαρντίν είναι η, η την ενδιαφέρει πολύ το θέμα αυτό, το έχει παρακολουθήσει με πολύ μεγάλη επιμέλεια και λυπάται πολύ που δεν μπορούσε να είναι παρούσα. Αλλά έγινε ένας μεγάλος σεισμός στη Βόρεια Ιταλία και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να... Σήμερα το πρωί και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να έρθει. Λοιπόν, είναι θέμα που έχει να κάνει με τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε, αυτήν την, σε αυτόν τον οργανισμό. Θα πρέπει βεβαίω και να καταβάλουμε το σχετικό ε, τέλος ε, συμμετοχής, αλλά ταυτόχρονα κερδίζουμε από την ε, συνάντηση ε, με εκπροσώπους από το Σουδάν, τη Ζιμπάμπουε, το Ουσμπεκιστάν, που είναι μέλη τη οργάνωση αυτή, και έτσι μπορούμε να προαγάγουμε και τον πολιτικό διάλογο που θα πρέπει βέβαια το ταχύτερο δυνατό να εντατικοποιηθεί. το θέμα του πώς θα μας ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, τακτικά ασφαλώς, και βεβαίως και το ζήτημα του πώς θα συμμετάσχει σε αυτές τις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στον διεθνή αυτό οργανισμό του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα οποία πολλές φορές έχουμε είτε μέσα από γραπτές δηλώσεις είτε από ψηφίσματα προβάλλει, φερρυπίν, χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία, ε, στο χώρο ιδιαίτερα τη παγκόσμιας αγορά του Φάμβακα, μεγάλη πτυτικότητα των τιμών που έχει καταγραφεί, διαφάνεια αγορά Είναι όλα αυτά θέματα τα οποία πιστεύουμε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο διάλογο και πάνω απ' όλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι και μέλη της ε, οργάνωσης αυτής μπορούν ε, να αφήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα εκπροσωπεί ω μία ενότητα, δεδομένου ότι πρόκειται για θέματα αρμοδιότητα, στο βαθμό μάλλον πρόκειται για θέματα αρμοδιότητα Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό προτείνει η κυρία Μουσκαρντίνη, την ενδιαφέρει ιδιαίτερα όπω είπα. Λυπάται ιδιαίτερα που δεν μπορούσε να είναι παρούσα εδώ, αλλά περιμένει να ακούσει τι προτάσει σα, συστάσει σα, υποδείξει σα, τι οποίε θα καταγράψω εγώ και θα, σας τις, διαβιβα... θα, θα τις, τις διαβιβάσω. Και ευχαριστώ πολύ του ευχαριστώ τους συναδέλφου. Θα ήθελα να στήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη που απουσιάζει η κυρία Μουσκαρδίνη. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση του θέματος. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους προσκεκλημένους μας, την κυρία Ινα Γκρόμαν, που είναι σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας, εξ ονόματος της ΙΚΑΚ για τον κύριο Τσεβέρνη που είναι πρόεδρος της Επιτροπής για τη Διεθνή Συνεργασία ανάμεσα στους ε, οργανώσεις Βάμβακος. Καλώς ορίσατε καταρχήν, σας ευχαριστούμε που ήρθατε και συνεργάζεστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μας διαφωτίσετε για τα πλανεκτήματα και τα κόστη Τη προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Πάμβακο. Κύρια Γκρόνμαν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίε και κύριοι, πριν να ξεκινήσω αυτή την παρουσίαση, για την εργασία της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος, ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν μιλώ εξ ονόματος της γερμανικής κυβέρνησης σήμερα, ούτε εξ ονόματος του Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας μου, ε, για το οποίο εργάζομαι, αλλά εξ ονόματος της ΣΥΚΑ και του διευθυντή της, του κ. Τέρι Τάουνσεν, που δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρόν. Λόγω άλλων ανελημμένων υποχρεώσεων έπρεπε να μιλήσει στην ΦΑΟ, στην Επιτροπή Οικονομικών και γι' αυτό και μου ζήτησε να κάνω τη δική του παρουσίαση. Εγώ, όπως σας είπα, εργάζομαι στο Υπουργείο Οικονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας και ασχολούμαι με τα διεθνή συμβουλευτικά όργανα για διάφορα αγαθά και παρακολουθώ τακτικές συνελεύσεις της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση για το παγκόσμια βιομηχανία Βάμβακος καλλιεργείται βαμβάκι σε 100 χώρες και παραπάνω. Είναι ε, μια από τις πιο σημαντικές καλλιέργειες όσον αφορά την χρήση της ε, γης μετά από την κράμβη και την σόγια. Ε, και μάλιστα 50 χώρες ασχολούνται με τις εξαγωγές και εισαγωγές βάμβακος πάνω από 100 εκατομμύρια οικογένειες ασχολούνται άμεσα με την παραγωγή βάμπακος. Όταν εξετάζουμε την οικογενειακή εργασία και τους εργαζόμενους στις παράπλευρες επιχειρήσεις όπως ας πούμε η μεταφορά και η αποθήκευση, μιλάμε για 200 εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με τον τομέα βάμβακος. Επίσης το βαμβάκι παρέχει απασχόληση σε παραπάνω εκατομμύρια για, σε, σε, κόσμο δηλαδή που εργάζεται στη γεωργική βιομηχανία, στα λοιπάσματα, στην υφαντουργία και ούτω καθεξής. Η καλλιέργεια βάμβακους ε, βελτιώνει την ασφάλεια σε τρόφιμα, την ε, συνθήκες διαβίωσης ανθρώπων ε, στις Νασία, στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική. Είναι μεγάλος παράγοντας πλούτου. 60 δις εκτιμάται ότι είναι η αξία του βάμβακος φέτος μόνο. Και βεβαίως αυτός ο όγκος ε, αιτιολογεί το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων και την ανάμειξη των κυβερνήσεων στην, στο βαμβάκι. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές από 7 εκατομμύρια τόνους το 1950 και 51 σε 27 εκατομμύρια τόνους τώρα. Από το 1950 ο μέσος όρος ανάπτυξης της παραγωγής βάμβακος ήταν 2,5% ετησίως. Νέες τεχνολογίες, πιο εκτεταμένη χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών και νέες ε, περιοχές ε, όπου καλλιεργείται το βαμβάκι οδήγησαν σε αυτές τις αλλαγές στην παραγωγή. Η παγκόσμια παραγωγή έχει αυξηθεί από τα 200 κιλά ανά εκτάριο στα 750 ε, κιλά ανά βιοτεχνολογία, βελτιωμένη άρδευση, στοχευμένες εφαρμογές ζανιοκτώνων, βελτιωμένη χρήση των ε, λιπασμάτων και η διαχείριση των ε, καλλιεργειών οδήγησαν σε μεγαλύτερο χαμηλότερο κόστος αυτής. Από τη διάρκεια της δεκαετίας 70, 80 και 90 η μέση τιμή ε, που δινόταν στα, δινόταν στα ήταν κάτω από το κόστος ε, παραγωγής για πολλούς καλλιεργητές ε, και για πολλά χρόνια. Πολλές χώρε χώρες παραγωγή ανταποκρίθηκαν δίνονταν επιδοτήσεις. Ε, η προσαρμογή γρήγορη μάλλον της βιοτεχνολογίας το 2000 οδήγησε στην... στο να αναπτυχθεί η προμήθεια γρηγορότερα από τη ζήτωση. Έξι Αναλύβρα. Τα, οι μέσες τιμές ε, για το βαμβάκι αναμένονται να είναι 80 σέντς με ένα δολάριο ανά λίβρα αυτήν την ε, δεκαετία. Το κόστος της παραγωγής ε, φτάνει κατά μέσο όρο τα 55 σέντς ανά λίβρα. Άρα λοιπόν θα είναι πιο κερδοφόρια η καλλιέργεια βάμβακος ε, φέτο, ε, μάλλον αυτή τη δεκαετία από ό,τι τις προηγούμενες δεκαετίες που σας ανέφερα. Και να δούμε μια εικόνα της εργασίας της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ΑΕΚΑΚ είναι ένας, ένας, μια ένωση σε 22 χωρών που παράγουν βαμβάκι. Το 39 Ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός, ο ετήσιος προϋπολογισμός είναι 2 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία το 85% προέρχονται από τις επιδοτήσεις των των κυβερνήσεων και το υπόλοιπο από συνδρομές και συμμετοχή των, σε διάφορα σεμινάρια. Η γραμματεία αποτελείται από 11 μέλη που αντιπροσωπεύουν 10 χώρες. Η ΆΕΚΑΚ δημοσιεύει τα έγγραφά της στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά ε, μηνιαίως και σύνοψη αυτών υπάρχει στα ρωσικά και στα αραβικά. Αποστολή της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής Βάμβακος είναι να βοηθήσει τις κυβερνήσεις όσον αφορά την εξυγίανση της οικονομίας του βάμβακος ε, μέσω της διαφάνειας, μέσω, χρησιμεύει επίσης ως εκαθαριστικός ε, οίκος, ε, καθώς και για τα, ως βήμα για συζήτηση θεμάτων διεθνούς σημασίας. Δίνει πληροφορίες σε σχέση με την επίλυση των προβλημάτων, προωθεί την συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων, και αποτελεί έναν αντικειμενικό στατιστικό παρατηρητή για τις χώρες που εμπορεύονται βαμβάκι. Παίζει έναν ε, μοναδικό ρόλο ως καταλήτης για επικοδομητική αλλαγή ποτέ δεν έπαιξε ρόλο στην θέσπιση των τιμών της αγοράς, ούτε παρενέβη στους μηχανισμούς της αγοράς. Ωστόσο, η Γραμματεία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που είναι επίκαιρες και ε, κέρυες για όλο όκληρο τον τομέα και αξιολογεί τις συνθήκες της αγοράς. Η ICAC είναι η πρώτη πηγή διεθνών δεδομένων για την ε, παγκόσμια βιομηχανία βάμβακος. Οι πληροφορίες που δίνονται από την ΑΕΚΑΚ είναι η χρήση, τιμές, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, μετρώνται οι προβλέψεις, μετρώνται οι προβλέψεις για την κατανάλωση και τη ζήτηση βάμβακο στον κόσμο αναπεριφέρεια και είναι και βασική πηγή για, στατική, για τις στατιστικές όσον αφορά τη ζήτηση ινών. Η γραμματεία εργάζεται ως ε, καθαριστικός οίκος για τεχνικές πληροφορίες, ούτως ώστε πάνω από 3.500 ε, ε, ερευνητέ διδακτορικού επίπεδου που ασχολούνται με την τεχνολογία βάμβακος να γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει. Έχουμε ερευνητικά προγράμματα καθώς και αιτήσια προγράμματα κατάρτισης για τους ερευνητές τόσο από χώρες παραγωγούς όσο και από χώρες καταναλωτές. Βοηθά επίσης στην χρηματοδότηση περιφερειακών σκέψεων ε, σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και κάνει δημοσιεύσεις για τις ε, πρακτικές παραγωγής, έτσι ώστε να ενημερώνεται ολόκληρη η ερευνητική κοινότητα βάμβακα. Μιλάμε για βιολογικές ε, καλλιέργειες ε, και ε, όχι μόνο. Εμείς συμμετέχουμε στην επίτευξη συνένεσης όσον αφορά τα πρότυπα ταξινόμησης που θέλουμε να αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα και έχει δημιουργηθεί και μια task force για την ε, ετυποποίηση. Η γραμματεία διευκολύνει επίσης τις προσπάθειες που θέλουν ε, να κάνουν κάποιες χώρες ε, για να αποφύγουν την μόλυνση του βάμβακα. Η ΆΕΚΑΚ αποτέλεσε καταλήτη επικοδομητικό για την ανταπόκριση της παραγωγής και της κατεργασίας του Βάμβακος από το 1990 και έπειτα και δίνει πληροφορίες στις χώρες που θέλουν ε, να εξαλείψουν ε, τις ε, κοινωνικές επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις, αλλά και προωθώντα τι καλύτερε προοπτικέ. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για τι κοινωνικέ, οικονομικέ και περιβαλλοντικέ ε, επιπτώσει του βάμβακο δημιουργήθηκε το 2006. Συμπεριλαμβάνει εμπειρογνώμονε για διάφορε πτυχέ τη παραγωγή βάμβακο και τη κατεργασία αυτού. Ρόλο τη είναι να δίνει πληροφορίε, να κάνει ρεαλιστικέ συστάσει για τη βελτίωση σε διαβούλευση με άλλου διεθνεί οργανισμού όπω ε, ο Διεθνή Οργανισμό Υγεία και η ΦΑΟ και Επίσης έχουμε, ε, μάλλον ο ΙΚΑΟ εκδίδει διάφορες εκθέσεις όσον αφορά τις κοινωνικές επιπτώσεις παραγωγής βάμβακος, τα συστατικά του εργατικού κόστους για την παραγωγή βάμβακος, η χρήση ενέργειας, η χρήση ζανιοκτώνων στο βάμβακα στις μεγάλες χώρες παραγωγούς και όλες αυτές οι εκθέσεις υπάρχουν στο site του ICAC. Η ICAC γνωρίζεται στην, στο Διεθνές Ταμείο Αγαθών. 22 προγράμματα για το ΒΑΜΒΑΚΑ υποβλήθηκαν από τον και που αξιολογήθηκαν στη, προς 17 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα προγράμματα υποστηρίχθηκαν από το Ταμείο. Έχουμε επίσης, λειτουργούμε ως βήμα για τη συζήτηση διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την βιομηχανία βάμβακος και δίνουμε ευκαιρίες ώστε να υπάρξουν διαβουλεύσεις για θέματα αμοιβαίων ενδιαφέροντος μεταξύ χωρών παραγωγών και χωρών καταναλωτών βάμβακος. Από πρόσφατες συνεδριάσεις η ΆΙΚΑΚ έχει εγκρίνει την μετακίνηση προς άλλες μεθόδους ελέγχου το βάμβακος. Έχουμε μιλήσει για τη χρήση της βιοτεχνολογίας, ε, ρίχθηκαν πολιτικές ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ΚΑΚ ε, συμβάλλει στην ασφάλεια τροφίμων. Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν ότι συγκεκριμένα ζανιοκτώνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγική βάμβακος και έπειτα οι χώρες συμφώνησαν ε, για να δίνουν τυποποιημένες στατιστικές για την παραγωγή βάμβακος έτσι ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια και να δοθούν και περισσότερες πληροφορίες ε, στους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων. Η ΆΕΚΑΚ ε, φέτος θα κάνει την 71η της Ολομέλεια ε, στην Ελβετία. Θέμα της φετινής Ολομέλειας είναι η βιωσιμότητα και η αλυσίδα αξίας του βάμβακος. Στόχος είναι να κατανοήσουμε τι σημαίνει ακριβώς βιωσιμότητα στην, για τη βιομηχανία βάμβακας τόσο στις χώρες κατανάλωσης όσο και στις χώρε χώρες ε, παραγωγής αλλά και στις αναπτυσσόμενες και λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαρίστως θα υποδεχτούμε και προσώπους της Ένωσης. Η ΚΑΚ ως ε, Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή για το Βαμβάκι παίζει ε, έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της βιομηχανίας βάμβακος. Ε, η... Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και χρήσιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος. Ε, έτσι ολοκληρώνεται η παρέμβασή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση του ρόλου και της αποστολής της ΆΙΚΑΚ. Να ακούσουμε τώρα τους ενδιαφερομένους, δηλαδή της ενώσεις ε, βαμβακοπαραγωγών, τον κύριο Ταβερνιέ, που είστε. Ναι κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Ήθελα απλώς να επισημάνω ένα-δυο πράγματα τα οποία συνέβησαν ε, τα τελευταία χρόνια. Για το 2010-2011 η Ινδία απαγορεύει τις εξαγωγές και ως αποτέλεσμα οι τιμές βάμβακος από 1,5 ευρώ ανέβηκαν στα 3,5 ευρώ. Αυτές οι κυβερνητικές δράσεις είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να αποφεύγονται και θα πρέπει να καταπολεμώνται. Γι' αυτό και φορείς όπως η Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος αποτελούν τον ιδανικό οργανισμό για να καταπολεμήσουμε τέτοια φαινόμενα. Φέτος και πάλι, δηλαδή για την εσοδεία 2011-2012, υπήρχε απαγόρευση για τις εξαγωγές και ως αποτέλεσμα οι τοπικές τιμές Βάμβακο στην Ινδία μειώθηκαν κατά 50% και η τοπική κλωστοϊφαντουργία μπορούσε να αγοράσει πολύ φθηνότερα, το, φθηνότερα τοπικά το βαμβάκι του από ότι η εταίροι του σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός και επομένως και πάλι φορείς όπως ο ΆΙΚΑΚ μπορούν να προωθήσουν θέματα αυτής της μορφής και μπορούν να τιμωρήσουν κυβερνήσεις οι οποίες αναλαμβάνουν τέτοιες ε, δράσεις. Ευχαριστώ. Let's open the... Καλώς. Ας ακούσουμε λοιπόν ερωτήσεις, σχόλια. Η κυρία Κέλλερ πρώτα. You'll be next. This is Thank you. Ναι, εσείς μετά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Στα όσα είπατε στο τέλος για την ε, αποτροπή περιορισμών ε, εξαγωγών, όπως είδαμε από την Ινδία, όπως που αναφέρατε. Πώς θα το καταφέρετε αυτό ακριβώς. Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Ναι, ναι, νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ίσως και άλλες ερωτήσεις. Ο Πρόεδρος. Ναι, έτσι, έτσι ήθεστε, ήθεστε εδώ. Ακόμα πρώτα αρκετές ερωτήσεις και μετά δίνουμε το λόγο στους ομιλητές μας. Ενημερωτική είναι αυτή. Έχετε και άλλη ερώτηση, μάλιστα. Η Επιτροπή Βάμβακος επικεντρώνεται περισσότερο στους παραγωγούς, χώρες παραγωγούς. Αλλά βλέπω και κάποιες ε, προσφυγές εις βάρος ε, Γερμανών, ε, Ευρωπαίων εισαγωγών από ένα γερμανικό δίκτυο δικαστικής αρρωγής για δραστηριότητες πολυεθνικών επιχειρήσεων κατά της Γερμανίας, Ισπανίας, Ελβετίας, Αγγλίας, Γαλλίας για παραβιάσεις των δικαιωμάτων, που δεν μερίμνησαν αυτές οι ε, επιχειρήσει να σεβαστούν. Και ρωτώ αν είστε ενήμεροι αυτών των προσφυγών και αν τις υποστηρίζετε στα σημεία, εθνικά σημεία επαφής του όσα ή ενδεχομένως να έχετε κάποια αντίστοιχα σημεία επαφής δικά σας πώς λειτουργούν, ποιος μπορεί να απευθυνθεί σε αυτά. Τι περιμένει λοιπόν η Επιτροπή και επίσης, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, πώς και σε ποιο βαθμό μπορεί να εμπλακεί σε τέτοιου είδους αποφάσεις του το Κοινοβούλιο. Ναι, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την κυρία Κρόμα για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Πρέπει να ομολογήσω ωστόσο ότι δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μα κάνει την παρουσίαση εκ μέρου τη Διεθνού ε, Συμβουλευτική Επιτροπή βάμβακο εκπρόσωπο του Γερμανικού Υπουργείου των Εξωτερικών τη. Μπορεί να μα δώσει εξηγήσει τη. Έχω τον κατάλογο των μελών τη Επιτροπή, Διεθνού Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακο εδώ. Και στην παρουσίαση πρόσεξα ότι είπατε 100 χώρες περίπου του κόσμου παράγουν βάμβακα. Αλλά η ΙΚΑΚ έχει μόνο 42 μέλη, η συμβουλευτική σας επιτροπή. 42 μέλη στα οποία περιλαμβάνεται και η Φινλανδία και η Γερμανία. Ε, δεν έχω υπόψη μου, είναι βαμβακοπαραγωγές χώρες. Αλλά εάν έχετε χώρες βαμβακοπαραγωγές που είναι που δεν είναι μέλη και έχετε χώρε μη βομβακοπαραγωγέ που είναι μέλη, μήπω θα μπορούσατε να μα δώσετε κάποιε εξηγήσει. Και κάτι άλλο. Πέραν τη κεντρικότητα κατά τα φαινόμενα που διαπιστώνω εγώ και διορθώστε με αναπατώμε. Η κεντρικότητα στην ε, ε στελέχωση των ε, μελών της ΙΚΑΚ. Βλέπω λοιπόν από τα 42 μέλη ότι είναι όλα εθνικά κράτη. Κατά τύχην δε και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης και της Γερμανίας που ανέφερα νωρίτερα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνω την εξή παρατήρηση, κρίσιμη παρατήρηση κρίσιμο επιχείρημα για οποιονδήποτε παρακολουθεί, ακούει, αλλά ιδίω για τα μέλη τη Επιτροπή μα που φαντάζομαι εκπροσωπούνται εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτο, δεν είναι εθνικό κράτο, δεν έχει νομική προσωπικότητα. Και πάνω απ' όλα δεν έχει και την νομο, νομιμοποίηση να είναι κράτος μέλος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τακτικά, συστηματικά τέτοια νομιμοποίηση να την διεκδικείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναγνωριστεί ως κράτος μέλος αν το επιδιώκεται. Αλλά Κυρίως όσον αφορά τα δημοψηφίσματα που είδαμε και για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα έγιναν δημοψηφίσματα στη Γαλλία και στην Ολλανδία δύο από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη και απέτυχαν θα πρέπει να σας πω ότι εξ ονόματος της ομάδας μου, την, τιμή, την, οποία, την ομάδα την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, είμαι πολύ επιφυλακτικός για αυτή την πρόταση, διότι μου φαίνεται ότι για άλλη μια φορά η Ευρωπαϊκή Άνεση αποπειράται παρανόμως και παρατύπως να ε, δρά ως κράτος μέλος, ε, όπως ε, το να ανήκει σε μία συμβουλευτική επιτροπή παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση και κανένας δεν τον εξουσιοδοτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Ο κύριο Κουτάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ως σκιώδης ογητή για την ομάδα μου, θα πρέπει να πω ότι από την πρώτη συζήτηση, από την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, που έγινε, υποστηρίζω την προσχώρησή μας σε αυτό τη Συμβουλευτική Επιτροπή, διότι θεωρώ ότι θα μπορούμε να μιλούμε με μία φωνή. Θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την ίδια πολιτική για το βαμβάκι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως είπε και ο Τανιέλ Γκασπαρή, θα ε, προσδώσουμε και μεγαλύτερη βαρύτητα στο συγκεκριμένο κλάδο. Όσο δε ε, την αποστολή της συμβουλευτικής αυτής επιτροπής, ε, στόχος της είναι να υποστηρίζει κυβερνήσεις να προάγουν μια υγιή οικονομία βάμβακος παγκοσμίως ενώ ταυτόχρονα ε, θα πρέπει να υπάρχει και διαφάνεια για την παγκόσμια βαμβακοπαραγωγή. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ε, ενταχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την Συμβουλευτική Επιτροπή θα μπορούμε πραγματικά να επηρεάσουμε τις χώρες οι οποίες εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται παιδιά, που χρησιμοποιούν την παιδική εργασία για, ε, για την παραγωγή βάμβακος. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να πιστούν οι χώρες αυτές να σταματήσουν τις πρακτικές τους. Συνεπώς, θα ήθελα να θέσω και μία ερώτηση προς τους εκπροσώπους της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένουμε προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για το θέμα αυτό. Πόσο πρέπει να περιμένουμε προκειμένου να υπάρχει μια, ένα θεματολόγιο το οποίο θα απαγορεύει την ε, εκμετάλλευση των παιδιών μέσω παιδικής εργασίας και να υπάρχει συγκεκριμένη σύσταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρε. Ανήκουμε και σε... Ανήκουμε και σε άλλους διεθνείς οργανώσεις προϊόντων, επομένως δεν είναι μόνο αυτή που μας αφορά. Επιπλέον, η εμπορική πολιτική είναι πλέον αποκλειστική αρμοδιότητα και θα πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε σε τέτοιους διεθνείς οργανισμούς προϊόντων, ώστε να μπορούμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ρούμαν. η οποία μας είπε ότι είναι εκπρόσωπος της ICAG και δικαίως και όχι της γερμανικής κυβέρνησης. Η ICAG αποτελείται από αρκετέ χώρες και δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει ότι έχουμε κάποιον ο οποίος ε, μπορεί να έχει μια διπλή ιδιότητα. Ανήκει ε, στην κυβέρνηση μιας χώρας, είναι υπάλληλο μιας χώρας και ταυτόχρονα εργάζεται και για την ΕΚΑΚ. Κυρία Ρόμεν, έχετε το λόγο να απαντήσετε στις ερωτήσεις και να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και για τις διευκρινήσεις. Όπως είπα, δεν εκπροσωπώ τη γερμανική κυβέρνηση Προσπάθησα να το διευκρινίσω. Αλλά δεν έχουμε κανένα από την Συμβουλευτική Επιτροπή α, Βάμβακος. Και επειδή γνωρίζω κάπως το έργο της ΑΙΚΑΚ, παραλάβα εγώ το λόγο και συμφώνησα να έρθω συνεδρίαση, γιατί δυστυχώς την τελευταία στιγμή ανακοινώθηκε αυτή η αναγκαία παρουσία της ΑΙΚΑΚ. Αναφερθήκατε στα παράπονα μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα εθνικά σημεία επαφή ε, του ΟΣΑ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν θεσμοθετημένες σχέσεις μεταξύ των ε, σημείων επαφής του ΟΣΑ και της ε, Οριζόντιας Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η ΆΙΚΑΚ ασχολήθηκε με το θέμα της παιδικής εργασίας στη Συλλογή Βάβακος Μάλιστα αποτέλεσε το επίκεντρο δύο συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής της ΑΙΚΑΚ το 2008 και το 2009. Εκεί εκπρόσωποι από το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, από τη UNICEF και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας ε, προσκλήθηκαν. Μάλιστα έγινε ένα σεμινάριο για τις βέλτιστες πρακτικές από την ΆΙΚΑΚ για να χρησιμοποιούνται υπεύθυνε πρακτικές ε, σε όλη την αλυσίδα εκμετάλλευσης βάμβακος και να αποφευθεί η προσφυγή σε παιδική εργασία. Έτσι γίνεται μια προσπάθεια φύπνισης πρόθεσης του διαλόγου για το θέμα αυτό, της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας. Δεν έχει κανονιστική ισχύ. Υπάρχει και ένα πάνελ για το κοινωνικό περιβάλλον και τις οικονομικές επιδόσεις της βιομηχανίας Βάμβακος και στην Επιτροπή αυτή αναφέρθηκε το ζήτημα αυτό, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για την παιδική εργασία που αποτέλεσε θέμα της ημερήσιας διάταξης σε όλες τις ολομέλειες από το 2009. Επίσης, το θέμα της βιωσιμότητας ασχολεί την Ολομέλεια και η αποφυγή της ε, παιδικής εργασίας είναι ένα από τα σημαντικά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην ΆΙΚΑΚ μη βαβακοπαραγωγών χωρών. Η ΆΙΚΑΚ δεν είναι οργανισμός βαβακοπαραγωγών χωρών, γιατί συμμετέχουν εκεί και εμπορικές ε, οργανώσεις διανομής ε. συμμετέχουν σε αυτό το φόρουμ συζήτησης. Είναι σημαντικό λοιπόν για τη βιομηχανία ακόμη ε, και μη βαβακοπαραγωγών χωρών να συμμετέχει στην ΆΙΚΑΚ. Αυτά προς το παρόν. Θα ήθελα να πω ότι αυτό ισχύει για, όλα, για όλες τις διεθνείς οργανώσεις ε, διαφόρων προϊόντων. Γιατί εκεί συμμετέχουν και καταναλωτές, έμποροι, χρήστες και όχι μόνο παραγωγή. Το ίδιο ισχύει και στο κακάο, μια πρόσφατη περίπτωση που μας απασχόλησε. Λογικό είναι να ισχύει και στο βαμβάκι. Ο κύριος Σταβερνιέ τώρα. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που σας απίθυναν τα μέλη της Επιτροπής ή έχετε κάποια σχόλια. Καταρχήν, απαγόρευση ε, εξαγωγών από την Ινδία, δεν κάνω λάθος. Η Ινδία ήταν μέλος της ΑΙΚΑΚ, οπότε μέσω ε, της συμβουλευτικής αυτής επιτροπής μπορούμε να ασκήσουμε πιέσεις και ε, να κάνουμε διαβήματα στα διάφορα Ινδικά υπουργεία για να αναλυφθούν δράσεις και μέχρι στιγμής είχαμε αρκετά θετικά αποτελέσματα γιατί πριν από τρεις εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, καταργήθηκε αυτή η απαγόρευση. Έτσι συνήθως λειτουργούμε. Καλώς. Ποιος θα μιλήσει τώρα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής? Ο κύριος Μούζη. Έχετε το λόγο αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μία ερώτηση απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερη ερώτηση. Πόσο θα κοστίσει η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακο στην ΆΙΚΑΚ και ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία από την προσχώρηση στην ΆΙΚΑΚ. Ονομάζομαι Μάθιο Κις και εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο συχνή ερώτηση είναι τι περιμένουμε από την Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Βάβακο στην ΆΕΚΑ και για ποιο λόγο έχει νόημα η συμμετοχή μας εκεί. Να σας ενημερώσω και ως προς τις εξελίξεις ό,τι αφορά τη, τη συμμετοχή μας. Δεν είμαστε ακόμη μέλη, εξετάζουμε τη συμμετοχή μας, την προσχώρησή μας στην ΆΕΚΑ, αλλά δεν είμαστε ακόμη μέλη της ε, Συμβουλευτικής αυτής Επιτροπής. Συνεχίζονται οι συζητήσεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την προσχώρηση στην ΆΕΚΑΚ και μάλιστα ε, στη συνεδρίαση του Ιουνίου της ε, ομάδας προϊόντα του Συμβουλίου θα γίνει σχετική συζήτηση. Και μάλιστα το ακριβέ ζήτημα που υπάρχει σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στην οργάνωση αυτή είναι το θέμα τη συμβολή Ευρωπαϊκή Ένωση, τη συνεισφορά τη. Δεν έχει καθοριστεί ακόμη το ύψο τη συνεισφορά, τη εισφορά. Γιατί όταν θα προσχωρήσουμε στην ε, ΆΙΚΑΚ θα ενταχθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, θα καταβάλουμε μία μόνο εισφορά, όχι 27 διαφορετικές αλλά το ύψος αυτής της εισφοράς δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Επίσης θα πρέπει να, να καθοριστεί σε σχέση και με τις εισφορές των εννέα μεμονωμένων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλλον θα είναι χαμηλότερο από το άθροισμα των εννέα αυτών εισφορών. Γιατί, επαναλαμβάνω, θα είναι μία η θέση μέλους και άρα μία εισφορά. θα είναι γύρω στα 2 με 3 χιλιάδες ευρώ για άλλες περιφέρειες. Με άλλα μέλη πληρώνουν από μερικές εκατοντάδες μέχρι και ένα μέχρι και ένα εκατομμύριο ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει όμως ήδη σε, σε διοικητικά συμβούλια άλλων προϊόντων. Τώρα σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία θα έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για εμπόριο σε θέματα αυτά γιατί υπάρχει αποκλειστική κοινοτική αρμοδιότητα στου τομεί αυτούς. Επίση, θα καθόμαστε στην ίδια τράπεζα διαπραγματεύσεων με τους βασικούς εταίρους, τους παραγωγούς, τους εμπόρους, τους καταναλωτές. Οπότε θα ακούγεται η φωνή μας στον τομέα του βάμβακος και μάλιστα θα ακούγεται η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωση. Ω ενιαία φωνή. Επίση θα ήθελα να επισημάνω ή μάλλον να ολοκληρώσω αυτό το θέμα της συμμετοχής μας στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ε, ΕΚΑΚ και το θέμα της συμμετοχής της ανάμειξης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θέμα είναι μόλις δοθεί η έγκριση από το Συμβούλιο να ζητηθεί η γνώμη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΚΑΚ, γιατί έτσι ισχύει και για τις άλλες συμβουλευτικές επιτροπές προϊόντων. Πάντως, καλό θα ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη ό,τι αφορά την ανάπτυξη αρρωγής στον τομέα του βάμβακος είναι πολύ σημαντική και η στήριξη των κρατών μελών. Η συνολική πάντως ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Επιτροπής των Κρατών Μελών, ανέρχεται σε 300 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια στον τομέα του βάμβακος και εκεί θα είναι έντονη και προστιθέμενη αξία λόγω της συμμετοχής μας ε, στην οργάνωση αυτή. Γιατί έτσι θα προωθήσουμε και τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που μας ενδιαφέρουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ε, εξασφάλιση του επισητιστικού ανεφοδιασμού, το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχουν πολλοί τομείς που ξεπερνούν τον αμυγή εμπορικό τομέα. Γι' αυτό και είναι ενδιαφέρουσα η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τέτοια συμβουλευτική επιτροπή, όπως είναι η ΆΙΚΑΚ. Επίσης θα αξιολογηθεί η υποστήριξη προσφέρουμε σε διάφορα άλλα προϊόντα στις χώρες ΑΚΕ. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η αξιολόγηση και για τον τομέα του βάμβακος, γιατί είδαμε, αποτιμήσαμε τις προσπάθειές μας και ακριβώς επειδή έχουμε πολύ καλές επιδόσεις στον τομέα του βάμβακος, είμαστε και αξιόπιστος ε, εταίρος και παράγων σε αυτό το θέμα. Όπως αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο της ε, ΙΚΑΚ, είναι κάτι που το εκτιμά ιδιαίτερος και η ΆΙΚΑΚ και θα το επιδιώξουμε και περαιτέρω στο μέλλον. Νομίζω ότι απάντησα στι ερωτήσει που ακούσαμε. Αν υπάρχουν και συμπληρωματικές, πολύ ευχαρίστω να επανέλθω. Να δώσουμε λοιπόν και πάλι το λόγο στον κύριο Κασπαρή για να ολοκληρώσει τη συζήτηση. Έχετε κάτι άλλο να σχολιάσετε. Εν ονόματι της εισηγητρίας μπορώ να ευχαριστήσω για τις επιπρόσθετες πληροφορίες που μας δώσατε και φαντάζομαι ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία και να επανέλθει το θέμα σε μια άλλη ημερομηνία στην Επιτροπή αυτή προς περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ και τώρα έχουμε την εξέταση του σχεδίου εξέσεως στη συνεδρίαση 21 με ε, ε, ε, Ιουνίου οπότε χαιρετώ και αποχαιρετώ τους φιλοξενούμενους μας και περνάμε στο σημείο 15 πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις συνέπειες της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Δέρματος. Ο μιλήτρια είναι η κυρία Μουσκαρντίνη, είναι μια γνωμοδότηση υπομορφής επιστολής και η ουσία περιλαμβάνεται στην επιστολή που συνέταξε η κυρία Μουσκαρδίνη. Έχετε το κείμενο εις το φάκελό σας και αν δεν έχετε αντίδραση θα την στείλει ο πρόεδρος Σούλτ στα άλλα θεσμικά όργανα. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον κύριο Κάσπαρη σχετικά με το θέμα αυτό δηλαδή για την εξέταση του σχεδίου ψηφίσματος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η κυρία Μουσκαντίνη πριν από λίγο καιρό, σύμφωνα με το άρθρο 120 του εσωτερικού κανονισμού, έκανε ένα σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με ε, την ε, ε, κατάσταση στον τομέα της βυσοδεψίας, και είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πληγεί πολύ από την κρίση και ένας κλάδος ο οποίος έχει πάνω από 3.000 ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50.000 άτομα και έχει ένα τζίρο 10,7 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν είναι αμεληταίο. Υπάρχει έλλειψη πρώτων υλών. Αυτή αυτή στιγμή δεν είναι εύκολο να, ε, βρει κανείς δέρματα βυσοδεψίας. Οι τιμές είχαν μεγάλες ε, ε, αυξομοιώσεις, πράγμα το οποίο επηρέασε την τιμή στην αγορά. Υπάρχουν και άλλες τρευλώσεις της αγοράς λόγω περιορισμού εισαγωγών και επιπρόσθετους δασμούς που δεν συνάδουν με τους κανόνες Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επιπλέον το κόστος επεξεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι αλλού και π.χ. υπάρχουν και παρελκόμενα έξοδα όπως ο καθαρισμός των ε, βρώμικων υδάτων διότι εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν καθαρίζονται τα βρώμικα υδάτα απλώς διοχετεύονται κάπου αλλού. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε η επιστολή αυτή να μεταδοθεί και στα δύο άλλα θεσμικά όργανα για να δούμε αν, είναι, αν υπάρχει κάποια αντίδραση ή αν θα το ξανασυζητήσουμε διότι πρόκειται ε, για μια συγκεκριμένη βιομηχανία τον τομέα της βυρσοδεξίας αλλά ε, θεωρήθηκε ότι είναι σκόπιμο να πούν τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι κλάδοι της βιομηχανίας που είναι ίσως ειδικά θέματα αλλά στη σημερινή κρίση χρήζουν παρακολουθήσεων και γι' αυτό συμφωνήσαμε με την, Ευρωπα... με την εισηγήτρια να ζητήσουμε να στηριχθεί από την Επιτροπή μας αυτή η ενέργεια. Σας ευχαριστώ. Ήταν νομίζω όλα σαφή. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που έχει κάποιο σχόλιο. Ωραία, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κρέινοκ. Έχετε το λόγο. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν έχω τίποτα να σχολιάσω. Εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις μπορώ κάλλιστα να απαντήσω, αλλά δεν σχόλιο από πλευρά. Έχουμε λοιπόν κοινή συζήτηση για δύο ε, νομοθετικούς φακέλους που έχουν ως επί της ουσίας αρμόδια επιτροπή την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εμείς απλώς γνωμοδοτούμε. Καταρχάς για το μέσο για συνεργασία με τρίτες χώρες. Ε, ανήκε σε εμά, αλλά μας το στερήσανε και μετά έχουμε το 17 για τους κοινούς κανόνε και διαδικασίες για την εφαρμογή ε, των μηχανισμών για την εξωτερική δράση. Αυτή είναι εγκάρσια νομοθετική διαδικασία. Ο συντάκτη και των δύο γνωμοδοτήσεων είναι η συνάδελφο Σαντρικίενε από το ΕΛΚ, στην οποία δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή μας ε, πρέπει να γνωμοδοτήσει για την ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει ένα μηχανισμό εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Όπως θα θυμάστε, αυτή η έκθεση είχε ανατεθεί στην Επιτροπή μας ως αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αμφισβήτησε όμως την αρμοδιότητα της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου για τη συγκεκριμένη νομοθετική έκθεση και η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών αποφάσισε ότι λόγω της ίσης κατανομής ε, των Επιτροπών και βάση ε, των θεμάτων αυτών η αρμοδιότητα ε, της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου είναι στο άρθρο 1, παράγραφος 2, σημείο Β. Ενώ τα υπόλοιπα είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ε, δεν μπορεί να αλλάξει τα θέματα η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Η γνωμοδότησή μας λοιπόν βάση, γίνεται βάση του κανόνα 50 του κανονισμού. ο μηχανισμός εταιρικής ε, σχέσης. Να σας πω δύο λόγια για τον μηχανισμό αυτόν. Είναι μία από τις ε, πολιτικές εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουμε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ ε, που σημαίνει ότι έχουμε 116 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τη δράση αυτή. Τώρα, η συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προκύπτουν από την διμερή συνεργασία και γίνονται ενδιαφέροντε εταίροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπω είναι η Κίνα, η Ρωσία, χώρε τη Λατινική Αμερική και ούτω καθεξή. Στόχο είναι να προωθήσουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουμε τι μεγάλε παγκόσμιες προκλήσει σε συνδυασμό με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και ο κανονισμό αυτό θα αντικαταστήσει το χρηματοοικονομικό μέσο για τη συνεργασία, το ICI και το ICI-SIN, που ε, ολοκληρώνεται το 2013. Αλλά ε, το μέσο ευρωπαϊκής γειτονίας, ε, το προενταξιακό μέσο βοήθειας, καθώς επίσης ε, και τα νέα μέσα ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης θα συνεχιστούν και για την περίοδο 2014-2020. Το συναλλικό ποσό που προτείνεται για αυτές τις εξωτερικές σχέσεις είναι 56 δισεκατομμύρια ευρώ για το νέο δημοσιονομικό πολιτές πλαίσιο 14 εκατομμύρια για το IPA, για το μέσο γειτονία 20 ε, εκατομμύρια, 23 ε, εκατομμύρια και για το μέσο εταιρικής ε, σχέσης τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι η θέση μου, εξ όσων κατανοώ εγώ, είναι ότι οι πτυχές διεθνούς εμπορίου στο κανονισμό αυτό είναι ευρύτερες του ενός άρθρου το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού, οι περιοχέ παρέμβασης, ε, τα μέτρα εφαρμογή ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι η βασική αρχή για την επιτυχία αυτών των στόχων που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο που θέλουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και να δώσουν δυνατότητα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων για του Ευρωπαίου επιχειρηματίε. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω κάποιε τροπολογίε που πηγαίνουν πέραν τη αποκλειστική αρμοδιότητας τη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και ελπίζω ότι θα θεωρηθεί χρήσιμη συμβολή μα στου συναδέλφου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα συναντηθώ με τον εισηγητή, τον κύριο Μάριο Μάουρο, αύριο και ελπίζω να δεχτεί και να υποστηρίξει τις τροπολογίες που θα καταθέσω. Διότι ο στόχος μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κοινό, να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό αυτό το μέσο. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω 35 τροπολογίες και όλες αυτές ε, ε, ζητούν διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ε, και σε γενικές γραμμές σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο. Κάποιοι αφορούν το ICI, κάποιοι άλλοι αφορούν τις προηγούμενες ενδιάμεσες εκθέσεις για το ICI, το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη και ε, θεωρούμε ότι και οι δύο συνομοθέτες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχουν εξέσους στη στρατηγική διαδικασία και στη χάραξη της στρατηγικής μας και θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένοι τομείς συνεργασίας ε, και κάποιες ενδεικτικές ε, κατανομές των κονδυλίων θα πρέπει να είναι αντικείμενο των πράξεων και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και για την περίοδο 2014-2020, διότι αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κανονισμό και να καθορίζονται στο παράρτημα. Από εκεί και πέρα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει ε, εκτελεστικές πράξεις για να προχωρήσει τη, με την κατανομή των κονδυλίων. Μας ενδιαφέρουν επίσης και κάποιες άλλες πτυχές, διότι το, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να προάγει την διεθνή ανταγωνιστικότητα και να ε, καταπολεμά τον προστατευτισμό, να προάγει ε, νέε δυνατότητες για τους Ευρωπαίου επενδυτέ και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε μια τροπολογία προτείνω επίσης να μειωθεί το μερίδιο των ε, μη ουσιοδών τροποποιήσεων που γίνονται στα προγράμματα από το 20% στο 10%. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κρατήσει αυτό το μερίδιο στο 20% ε, είναι μια πρόταση που δεν μας βρίσκει σύμφωνος, διότι ε, είναι πολύ υψηλό αυτό το ποσοστό και δεν είναι πολύ σημαντικό για τα προγράμματα που έχουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέσο, αλλά θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό χρησιμοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων και να ακούσω και τις δικές σας τροπολογίες για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για την έκθεση. Όσον αφορά τώρα τους κοινούς κανόνες και τις διαδικασίες για την εφαρμογή των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική δράση, θα ήθελα απλώς να πω ότι προτείνω 19 τροπολογίες και ακολουθώ και πάλι την άγουσα που προτείνεται και στο μηχανισμό εταιρικής σχέσης. Εδώ ε, κάνω κάποιες μη ουσιαστικέ τροποποίησεις, ε, μείωση αυτών των μη ουσιαστικών τροποποίησεων από το 20% στο 10% για τους ίδιους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Προτείνω στο άρθρο 9 οι επιλέξιμες χώρες κυρίως οι αναπτυσμένες χώρες ε, να διαδραματίζουν προεξάρχοντα ρόλο στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές εμπόριο και να αντιμετωπίζουν παγκόσμιες προσκλήσεις και αυτό θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του κανονισμού κατά την άποψή μου. Για το άρθρο 16 τώρα προτείνω να είναι πιο σύντομη η ημερομηνία για τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση το αργότερο τον Ιούνιο του 2017 η ημερομηνία που προτείνεται είναι ακριβώς το μέσο της προγραμματικής περίοδου και αν δεν κάνω λάθος, η νωρίτερη αξιολόγηση της διαδικασία εφαρμογής και πιθανέ τροποποίησεις θα είναι προ όφελό μα, διότι θα έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο για να εφαρμοστούν οι αλλαγέ ε, στο υπόλοιπο μισό του προγράμματο για την πιο αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων προτείνω να προβλέπονται και τίσες εκθέσεις αξιολόγησης και όχι διετής όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά λοιπόν από πλευρά μου και προσβλέπω στις τροπολογίες σας μέχρι τις 12 το μεσημέρι της 1 η Ιουνίου. Δηλαδή εντός της εβδομάδος, την Παρασκευή το αργότερο και θα ψηφίσουμε στις 20 και 21 Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Ανδρικένα. Συζήτηση τώρα η κυρία Κέλλερ και πάλι. Ευχαριστώ. Έχω ένα γενικό σχόλιο. Αν έχουμε ένα χρηματοδοτικό μέσο που το αποκαλούμε μέσο εταιρική σχέση συνεργασίας με τρίτες χώρες, θα πρέπει να τονίσουμε την πτυχή της εταιρικής σχέσης, ε, τη συνεργασία δηλαδή. Και η πρόθεση στην προκογή των εμπορικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια λάθος εστίαση για ένα μέσο συνεργασίας. Γιατί όταν μιλούμε για συνεργασία έχουμε αμοιβέ συμφέροντα. Υπάρχει ένα δούνι και ένα λαβίν. Και αν πρόκειται για μέσο της εξωτερικής ε, πολιτικής, είναι μηχανισμός δράσης περισσότερο παρά μηχανισμός ικανοποίηση των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα ενδιαφέρει και η γνώμη των εταίρων μας και η εξυπηρέτηση των αμοιβαίων μας συμφερόντων. Ευχαριστώ. Δεν ζητά άλλο κανείς το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά την εισηγητριά μα για να δευτερολογήσει. Κυρία πέρε εκ μέρους Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προτιμώ να δώσω το λόγο στο συνάδελφο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τον Έλλης Μάθιους, γιατί έχουμε στενή συνεργασία μαζί του για το, για το μηχανισμό αυτό εταιρικής σχέσης. Ονομάζομαι Έλλης Μάθιους από την ΕΕΔ. Να πω λίγα λόγια σχολιάζοντας τις τροπολογίες της εισηγήτριας θα μιλήσω, θα απαντήσω γενικά, όχι τόσο διεξοδικά για τις τροπολογίες, προσπαθώντας να απαντήσω σε μερικές γενικές ερωτήσεις. Θεωρούμε ότι η βασική καινοτομία αυτού του πακέτου μέτρων που απαρτίζουν τον μηχανισμό με βάση το κεφάλαιο 4 της εξωτερικής ε, πολιτικής είναι κυρίως η, ο μηχανισμός εταιρικής σχέσης. Είναι περιορισμένο το γεωγραφικό πλαίσιο σχέση με το ισχύον ICI και το ICIC θα υποστηρίξει την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ένωσης όπως και τη στρατηγική του 2020. Γιατί μας ενδιαφέρει η ανταγωνιστικότητα, αλλά σε εταιρική σχέση, σε συνεργασία με τις άλλες χώρες του κόσμου για να αντιμετωπιστούν παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές, το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και το καθεξής. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που μέχρι στιγμή μα έλειπε από τι εξωτερικέ μα σχέσει. Και αυτό ο μηχανισμό καλύπτει ένα κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα μα επιτρέψει να ε, έχουμε σχέσεις με στρατηγικής σημασία για τα συμφέροντά μας χώρες. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα του κόσμου βέβαια, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρουν οι, οι βασικοί μας εταίροι όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ρωσία, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία. Με τι χώρε αυτέ είτε έχουμε ε, ε, συνεχείς, ε, συνεχιζόμενες οι εκκρεμείς εμπορικές συμφωνίες είτε προβλέπονται για το μέλλον τέτοιες εμπορικές συμφωνίες. Και προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τα αμοιβαία μας συμφέροντα. Δεν θα ξεκινήσουμε από τάβουλα ράζα σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα χρησιμοποιήσουμε τις συμφωνίες πλαίσιο που ήδη έχουμε συνάψει με τις χώρες αυτές, τα σχέδια δράσης που τα συνοδεύουν και θα χτίσουμε στα ήδη υπάρχοντα. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμος αυτός ο μηχανισμός και μεταξύ των τριών στόχων που έχουν προσδιοριστεί είναι και η εξωτερική, η διεθνής διάσταση της στρατηγικής του 2020, Ευρώπη 2020 και η παρουσία της Ένωσης ε, στο διεθνές προσκήνιο σε ό,τι αφορά τη διπλωματία της. Μας ενδιαφέρει η πρόσβαση στις αγορές και η ανάπτυξη επιχειρησιακών και εμπορικών ε, δυνατοτήτων ε, μέσω της εταιρική σχέσης και μέσω της προαγωγής των επιχειρήσεων αλλά και της ε, κανονιστικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Αυτό είναι θεμελιώδες αν ε, επιδιώκουμε κάποια σύγκληση των εταιρικών δραστηριοτήτων των εταίρων μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ένα πιο ασφαλές επιχειρησιακό περιβάλλον και επενδυτικό περιβάλλον. Αναφέρθηκε κάτι τέτοιο ακροθυγός. Βέβαια το ένα δισεκατομμύριο είναι μάλλον ε, ε, μικρό ποσό. Θα πρέπει να υπάρχει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων εξαιτία του σχετικά μικρού προϋπολογισμού και θα αξιοποιήσουμε και τη συμπληρωματικότητα για το ειδικό πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και θα φροντίσουμε να επιδιώξουμε συμπληρωματικότητα και συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Και υπάρχουν πολλές τροπολογίες που τονίζουν αυτή την ανάγκη συνέργειας και τη συμπληρωματικότητα. Είναι από αυτήν την άποψη πολύ εύστοχες τροπολογίες. Αυτά γενικά ως προς την πρόταση. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος από την ΔΕΦΚΟ θέλει να πει κάτι για το δεύτερο σημείο. Ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καταρχήν για τον κοινό εφαρμοστικό κανονισμό και τις δύο τροπολογίες. Στην πρώτη ζητάμε το σχέδιο γνωμοδότηση, το σχέδιο έκθεση να εξασφαλίσει μια ελαστικότητα, ένα περιθώριο λιγμών ως προς το 10-20% για την χρησιμοποίηση κάποιων κονδυλίων για ηλιμένες αποφάσεις και ηλιμένα μέτρα. Χαίρομαι για αυτό το περιθώριο λιγμών, μετά το 10% το 20% ως προς το ποσοστό, το ποσοστό είναι συζητήσιμο, αλλά η αρχή της ελαστικότητας μας βρίσκει σύμφωνος. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την διεύρυνση του κανονισμού σε χώρες που έχουν πολύ καλές επιδόσεις σε θέματα διακυβέρνησης, περιβάλλοντος κτλ. Καλή ιδέα, αλλά ποιος θα αποφασίσει ποιες είναι αυτές οι ενάρετες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα εφαρμογή εδώ. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις για το σχέδιο που προτείνατε, το σχέδιο γνωμοδότησης. Καλώς και επανερχόμαστε στην εισηγήτριά μας, την κυρία Αντρικιένα, για τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και όσους συνέβαλαν στη συζήτηση. Τώρα, για τα σχόλια που ακούσαμε, ο μηχανισμός αυτός προωθεί πρώτα απ' όλα τους στόχους και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Ταυτόχρονα όμως ο μηχανισμός αυτός θα επιδιώξει σαφή αποτελέσματα με βάση τους στόχους που θα έχουν συμφωνηθεί με τις τρίτες χώρες σε πολιτικό επίπεδο. Οπότε, ναι μεν έχουμε ως ζητούμενο την υλοποίηση των στόχων μας, αλλά θα γίνει και μια αξιολόγηση με διαφανή τρόπο με τους υπόλοιπους τέρους μας σε τοπικό ε, εθνικό, περιφερειακό επίπεδο και με τις κοινωνίες ε, των πολιτών αυτών των χωρών. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση ε, ως προς την επιδίωξη αυτών των στόχων. Πάντως θα το προσέξω και στις τραπολογίες. Θα συναντηθώ άλλωστε, όπως σας είπα σε λίγο, με τον αρμόδιο εισηγητή της Επιτροπής ΑΦΕΤ, τον κύριο Μάουρο, και θα το, το επισημάνω. καλή επιτυχία, καλή τύχη σας εύχομαι, αν θα πρέπει να το δείτε και με τον κύριο Μάουρο. Καλώς ολοκληρώσαμε τη κοινή συζήτηση για τα θέματα 16 και 17. Χρονοδιάγραμμα. 14 Ιουνίου λίγη η διορία και για τις διαγνωμοδοτήσεις. Α, συγγνώμη. 1η Ιουνίου. Λάθος στήλη κοίταζα. 1η Ιουνίου λίγη η ιουνιου λάθο στηλη κοιταζα 1 η ιουνιου λιγη η διορια για την κατάθεση τροπολογιών για τις δύο γνωμοδοτήσει. των σημείων 16 και 17. Αυτό μα το προανήγγειλε και η εισηγήτρια. Και έχουμε και μια ακόμη κοινή συζήτηση για άλλες δύο γνωμοδοτήσεις, σημεία 18 και 19, εξέταση του σχεδίου των σχεδίων γνωμοδότησης μάλλον που έχετε λάβει, αυτή τη φορά πρόκειται για γνωμοδοτήσεις που θα επιδώσουμε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων που είναι η αρμόδια κατ' ουσίαν. Δυστυχώς όμως απουσιάζει ο εισηγητή μα Δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Ας ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε. Για τα σημεία 18 και 19. η κυρία Σιμιώνοφ, η κυρία, ο κύριος Μισελ Κοσμίδης, η κυρία Μισελ Κοσμίδου, ε, ποια από τις δύο κυρίες. Είμαι η κυρία Σιμεώνοφ από την Δίζη Αγοράς, <clears throat> από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς, με συγχωρείτε, και είμαι στη διάθεσή σας αν με χρειάζεστε για κάτι. Ναι, έχουμε ένα σχέδιο γνωμοδοτήσεως οπότε μπορείτε να την, να την σχολιάσετε δεν, δεν χρειάζεται να ακούσετε τον εισηγητή διότι υπάρχει το κείμενο γραπτό Έχω διάφορα θέματα <clears throat> τα οποία θα ήθελα να αναφέρω και θα τα αναφέρω όλα μαζί διότι είναι ένα θέμα πολύ βασικό ε, και αναφέρεται και στις δύο προτάσεις η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενεργείας και ε, την σχετική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών διότι προβλέπεται μία επέκταση ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντίθετη στην ε, επέκταση της εμβελίας διότι αυτό που είναι βασικό αυτή τη στιγμή είναι να μην ε, ξεπεράσουμε το στόχο μας και να βρούμε μία συμβιβαστική θέση με το Συμβούλιο το οποίο έχει μία πιο συντηρητική προσέγγιση προβλέπεται και μία ρήτρα αναθεώρησης που μεταξύ άλλων αποβλέπει στην ε, αναθεώρηση άπαξ και εφαρμοστεί αυτό το μέσον διότι πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πιο βασικός τομέας ε, για τις τρίτες χώρες που κατά τη γνώμη μας ε, είναι συγκεκριμένες βιομηχανίες. Εάν δηλαδή το επεκτείνουμε δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλους τους τομείς κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προβλέπεται ένα καθεστώς διαφορετικό σήμερα με το οποίο θα πρέπει οι εκθέσεις να γίνονται κατά χώρα ενώ άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνονται κατά πρόγραμμα για να απαλληφθούν οι διαφορές μία επέκταση η οποία προβλέπει ότι κατά τη γνώμη του εισηγητή ε, θα πρέπει να δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί προσπαθεί να ισοσκελίσει τις προτάσεις αυτές και την καλή διακυβέρνηση ε, κατά τρόπον ώστε να καλυφθούν τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και η πληροφόρηση αυτή θα θέσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε επιχειρηματικό κίνδυνο ενώ από την άλλη πλευρά άλλες χώρες που δεν έχουν αναλάβει τα δραστικά μέτρα που προτείνουμε εδώ θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Ακόμη και, Ευρω... και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν υιοθετήσει τη σχετική νομοθεσία οπότε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος διαφοράς των διαφόρων καθεστώτων που θα ισχύσουν πράγμα το οποίο θα οδηγήσει σε μία ανάγκη για τις επιχειρήσεις να συμβιβάσουν ασυμβίβαστα στοιχεία και γι' αυτό θα προτιμούσαμε να υπάρξει κάποια ε, αμοιβαία αναγνώριση αργότερα στο μέλλον στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και κατά ε, προτίμηση θα έπρεπε να καλύψουμε τις διεθνείς προδιαγραφές και όχι αυτή τη στιγμή που θα απαιτήσουν πολύ πιο αυστηρές προϋποθέσεις από άλλες χώρες σε σχέση με την Ευρώπη. Ένα άλλος τομέας ο οποίος καλύπτεται είναι ε, το, η έκφραση συλλικής υποδομής που προβλέπει ότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε αυτή την πτυχή και θα πρέπει να απευθυνθούμε στι κυβερνήσεις τρίτων χωρών και όχι σε ορισμένες πλευρές οι οποίες θεωρούν ότι δεν έχουμε επιτύχει το στόχο μας και αυξήσει τη διαφάνεια διότι αυτό που μπορεί να είναι σημαντικό για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικό για τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε από τη θέση των τρίτων χωρών και να δούμε εάν μπορούν να υπάρξουν πληροφορίες σχετικά με τα χρήματα που θα πληρωθούν σε αυτές τις χώρες και να προσπαθούμε να δούμε ε, τι έγινε με τη χρηματοδότηση αυτή και αν έχουν κατανεμηθεί όπως θα έπρεπε θα έπρεπε. Τέλος έτσι θα καλυφθεί ένα κενό που ε, θα αποσαφηνίσει την κατάσταση και ε, θα αυξήσει και τη διαφάνεια επιτρέποντάς μας να επιτύχουμε το επίπεδο που επιζητούσαμε. Όσον αφορά την εξαίρεση. Έχουμε προβλέψει περιορισμένες εξαιρέσεις. Υπάρχει ένας κίνδυνος ε, για τους εργαζόμενους στην εταιρεία σε περίπτωση που υπάρχουν ποινικές ενέργειες, ποινικά αξιόπινες ενέργειες και αυτό είναι ευθύνη κρατών οι οποίες ε, δέχεται να ε, νομοθετήσουν προς αυτή την κατεύθυνση για να αποφύγουν τη διαφάνεια ενώ πιστεύουμε ότι οι ευθύνες είναι ευθύνες εταιριών και όχι μεμονωμένων εργαζομένων επιπλέον υπάρχει δυνατότητα βραχυπρόθεσμα να σκεφτούμε άλλες ε, ρήτρες grandfather clauses σχετικά με το τι χρειάζεται ε, να ε, προβλεφθεί για να μην υπάρχει περαιτέρω νομοθεσία σε τρίτες χώρες στα πλαίσια αυτής της γενικότερης ε, νομοθεσίας και κατά τα άλλα επιμένουμε στις προτάσεις που έχουμε διατυπώσει. Η κυρία Σαΐφη έχει ζητήσει το λόγο. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να πάρω το λόγο μετά τον κύριο Σόλτς διότι τώρα μόλις έφτασα και εγώ είμαι σκιώδης του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, επειδή τροποποίησαμε την ημερήσια διάταξη ήμουν ε, προετοιμασμένος ε, για το πρωί, γιατί δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω από την αρχή τη συνεδρίαση, όμως άλλη συνεδρίαση. Ευχαριστώ ε, την Επιτροπή για τις εξηγήσει και ευχαριστώ και την κυρία Σάιφη που, θα, που μου δίνει την ευκαιρία να αναφερθώ σε ένα άλλο ζήτημα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αρμόδια κατ' ουσία επιτροπή είναι η Επιτροπή Ανάπτυξης. Και Για άλλο θέμα μιλάει ο κύριος Σόλτς. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, λέει ο μιλητής. Για άλλη οδηγία πρόκειται. Μιλάμε για τα σημεία 18 και 19. Αρμόδια κατ' ουσία Επιτροπή είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Ναι, όντω, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι η αρμόδια κατ' ουσία Επιτροπή. Uh, Προσπαθούμε στην εγγνωμοδότησή μου να ακολουθήσουμε τη γραμμή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και προτείνουμε ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Δηλαδή δεν συμφωνώ με τις εξηγήσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βέβαια αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να συμβάσει κάπως τα πράγματα με τη θέση του Συμβουλίου, αλλά εμείς προσπαθούμε να ευθυγραμμιστούμε με τις επιμέρους επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις Επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης που ζητούν μια διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή. Γιατί ζητούμενο είναι η διαφάνεια. Όχι μόνο με τις αρχικές βιομηχανίες την εξορρεκτική δηλαδή, αλλά και τη δασοκομεία, τη γεωργία και άλλους τομείς. Θέλουμε και εκεί διαφάνεια. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη διαφάνεια σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα παρακαλώ να προσκαλέσω τους και ηγητές και από τις άλλες επιτροπές για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων και να αποφασίσουμε και την ακολουθητέα προσέγγιση για να γίνει ένας καλύτερος συντονισμός και να τηρήσουμε και το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και να προλάβουμε να ψηφίσουμε στη συνεδρίαση του Ιουνίου. Κυρία Σαΐφη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σόλτς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξηγήσει τους για ένα θέμα που είναι πολύ τεχνικό. Επί της ουσίας συμφωνώ. Θέλουμε περισσότερη διαφάνεια και νομίζω ότι όλοι θα βγούμε κερδισμένοι από μια ενίσχυση της διαφάνειας. Και αυτή την άποψη και οι δύο προτάσεις συνιστούν ουσιαστική πρόοδο. Σε ό,τι αφορά τους τρόπους εφαρμογής και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2004-109. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να υποβληθούν μερικές τροπολογίες και άλλωστε αντίστοιχες συζητήσεις ε, διεξάγονται σε όλες τις ε, επιτροπές που γνωμοδοτούν. Για παράδειγμα, θα πρέπει να διευκρινίσουμε την έννοια του σχεδίου στην οδηγία αυτή, του project. Θα καταθέσω μάλιστα και σχετική τροπολογία. και σε άλλα σημεία θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις και να συνεννοηθούμε με τον εισηγητή. Σε ό,τι αφορά την ε, επέκταση της ε, υποχρέωσης αναφοράς σε, όλες τις, ε, σε όλους τους κλάδους, δεν είμαι επιπισμένη για την πρόταση αυτή. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά την οδηγία στην εξωτερική και την δοσοκομική βιομηχανία, να αντλήσουμε απαραίτητα συμπεράσματα και μετά επ' ευκαιρία μιας αξιολόγησης τότε να κρίνουμε αν είναι σκόπιμη η επέκταση αυτής της υποχρέωσης αναφοράς και στους υπόλοιπους τομείς. Επίσης, ό,τι αφορά τις εξαιρέσεις ε, για τις επιχειρήσεις ε, που ασχολούνται με την ε, υλοτομία, είμαι επιφυλακτική. Πολύ φοβάμαι ότι θα χρησιμοποιήσουν την εξαίρεση αυτή πολλές επιχειρήσεις για να παρακάμψουν τις υποχρεώσεις τους. Προτιμώ μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση. Άλλωστε, πριν από μια αναθεώρηση θα πρέπει να γίνει η μελέτη και αξιολόγηση της κατάστασης. Αυτές είναι προς το παρόν οι παρατηρήσεις μου και θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τον εισηγητή. Για να επανέλθουμε τώρα στον συντάκτη των γνωμοδοτήσεων. Ακούσαμε τις ενστάσεις και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυρίας Σαΐφη για τις προτάσεις σας. Πέστε μας, ε, ε, προτείνετε να διευρυνθούν οι υποχρεώσεις για τις πληροφορίες. Μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα βεβαίως τις παρατηρήσεις. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο πτυχές προς τους συναδέλφους, διότι θεωρώ ότι σαφώς και πρέπει να δούμε σε ποιον τομέα πρέπει να επικεντρωθούμε. Προγραμματισμός, αναπρόγραμμα και αναχώρα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει για άλλη μια φορά να αρχίσουμε να συζητούμε για το κατά πόσον θα πρέπει ευθύ εξ αρχής να προσπαθήσουμε να έχουμε μια ευρύτερη προσέγγιση το οποίο είναι ακόμα υποσυζήτηση στις άλλες επιτροπές. Να έχουμε μια κοινή ε, προσέγγιση δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο αυτό το μητρό διαφάνειας. Και μέσω αυτού να εξετάσουμε πού βρίσκονται τα πραγματικά συμφέροντα των χωρών μελών, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διότι αυτές οι δύο διαφορετικές θέσεις που αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν μέχρι τούδε, θα μπορούσαν ίσως να δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε πραγματικά περισσότερη διαφάνεια στην αμοιβαία συνεργασία δημιουργία αμοιβαίων πλαισίων για να δραστηριοποιούνται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά να επικεντρωνόμαστε ταυτόχρονα και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε μελλοντική οδηγία. Ίσως όμως να είναι και μια ευκαιρία για να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο και να κάνουμε κάποιες ανταλλαγές απόψεων ε, μεταξύ των σχεδόν εισηγητών και εμού. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνω τη συζήτηση. Τώρα, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών η 1η Ιουνίου, 12 το μεσημέρι και για τις δύο γνωμοδοτήσεις. Με αυτό λοιπόν ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση. Επειδή δεν έχουμε αρκετό κόσμο, αναβάλλεται η ανακοίνωση. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9. Έχουμε αρκετά θέματα να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.